D'après. Do we say I reopen? Yeah. Uh, I, I, the, the sitting is resumed. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung ist wieder aufgenommen. Möchte nicht in die Tag. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, αρχίζει η συνεδρίαση. Δεν θέλω να μπούμε στην ημερήσια διάταξη. χωρίς να εκφράσουμε κι εμείς ε, τον αποτροπιασμό μας για την ε, βιότητα με την οποία δολοφονήθηκε χθε ε, ένας στρατιώτης της ΗΠΑ και θα παρακαλέσω τον Πρόεδρο να μεταφέρει την, τα συλληπιτήριά μας, τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Δεν συνηθίζεται να παίρνω το λόγο, αλλά έχω ένα ερώτημα που πρέπει να θέσω στους φίλους σοσιαλιστές. Έχει τελειώσει στη Βουλγαρία η προεκλογική εκστρατεία, τα αποτελέσματα είναι πλέον γνωστά. Ίσως να σχηματιστεί κυβέρνηση σήμερα, να υπάρξει κυβερνητική πλειοψηφία ε, και δεν αποκλείουν οι ε, ε, σοσιαλιστές την επίσημη ή ανεπίσημη στήριξη του κόμματος ΑΤΑΚΑ. Έτσι είπε ο εκπρόσωπός τους ότι θα πιούμε και αυτό το πικρό χάπι. Θέτω λοιπόν το ερώτημα στη σοσιαλιστική ομάδα. Είστε όμοιροι του Στάνισεφ, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Γιατί να καταπιείτε το χάπι της συνεργασίας με το ξενοφοβικό και ακροδεξιό κόμμα το οποίο απορρίπτει το ευρωπαϊκό μέλλον της Βουλγαρίας θεωρεί ότι οι Ευρωπαίοι πρέσβεις και επενδυτές είναι απικιοκράτες που οφείλουν να τους διώξουν από τη χώρα. Αυτή η διαδικασία δεν θα υπονομεύσει γενικότερα μια τέτοια κυβέρνηση στις σχέσεις της με την Ευρώπη ή μήπως για την περίπτωση αυτή υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Κατηγορείται τη μία κυβέρνηση για το τι κάνει κάτι και δεν κατηγορείται μία άλλη που κάνει το ίδιο. Κοιτάξτε, έχω εμπιστοσύνη εγώ σε εσά και θα πρέπει να δώσετε μια απάντηση. Ο συνάδελφος Σαλόμ. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Ντόλ καλά κάνει και εμπιστεύεται τη δημοκρατικότητα των σοσιαλιστών. Γιατί αναμφίβολα εμείς οι σοσιαλιστέ είμαστε η ομάδα, ίσως όχι η πιο μεγάλη, αλλά δεν είμαστε λιγότερο σημαντικοί από οποιαδήποτε πολιτική ομάδα και ανέκαθεν ήμασταν υπέρ της δημοκρατίας στην Ευρώπη για την οποία και παλεύουμε. Και επίσης δίνουμε για τη μάγια δημοκρατία και σε άλλες χώρες εκεί που υπάρχουν κάποιες κυβερνήσεις τις οποίες το λαϊκό κόμμα σέβεται και προστατεύει ακόμα και από αυτή να εδώ τη θέση από αυτό εδώ το ημικύκλιο. Λέει για ομοιρία ο κύριος Ντόλ, όχι εμείς. Εμείς δεν είμαστε. Εμείς απλώς υπηρετούμε τις ε, αρχές μας και τις αξίες μας. Thank you very much, President. Do you have any special Έχετε κάποιο πρόβλημα, είμαι, επειδή είμαι γυναίκα σας ενοχλεί που πήρα το λόγο. Κύριε Ντόλ, μπορείτε να φορέσετε τα ακουστικά σας. Σας ευχαριστώ που θέσατε το θέμα αυτό. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Σας σέβομαι να σας υπενθυμίσω να ακούγατε τις ίδιες παρατηρήσεις, να άκουγα τις ίδιες παρατηρήσεις όταν σχηματίσαμε εμείς μια κυβέρνηση, όταν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το αντίστοιχο βουλγαρικό, σχημάτισε μια κυβέρνηση πριν τέσσερα χρόνια στη Βουλγαρία με την υποστήριξη του ιδίου του ακραίου κόμματος, το οποίο τώρα αναφερθήκατε. Αγαπητοί συνάδελφοι, προβλέπετε ψηφοφορία ε, στην ημερησία διάταξη. Μπορούν όλοι να λάβουν το λόγο, οι πολιτικές ομάδες. Κυρία Χάρμς, αλλά μετά παρακαλώ να κλείσουμε τη συζήτηση. Κυρία Χάρμς. Αγαπητέ Γιώζεφ Ντάουλ, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι δεν είναι αμεληταίο το γεγονός ότι ο κύριος Ντάουλ έθιξε αυτό το θέμα σήμερα. Νομίζω όμως ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να ανησυχούμε μόνο για τη Βουλγαρία, όχι μόνο για τις δημοκρατικές εξελίξεις στη Βουλγαρία. Υπάρχει μια ολόκληρη σειρά κρατών όπου είναι όλο και πιο δύσκολο να εντοπίσει κανείς τις ευρωπαϊκές αξίες και την δημοκρατία. Τον προηγούμενο μήνα συζητήσαμε για την Ουγγαρία. Ε, παλαιότερα είχαμε ξανασυζητήσει για τη Ρουμανία και εκεί εξεπλάγησαν οι φιλελεύθεροι. Ε, πολύ καθυστερημένα συζητήσαμε για την Ιταλία. Πολύ πιθανό λόγω των εξελίξεων στην Ελλάδα, λόγω της χρυσή αυγή, θα κληθούμε σύντομα να συζητήσουμε για την Ελλάδα. Εδώ λοιπόν δράτω με τις ευκαιρίες και θέλω να σας πω ότι η έκθεση Ταβάρες, λόγω της συζήτησης που γίνεται στην Ουγγαρία, η έκθεση αυτή απαριθμεί ένα, περιλαμβάνει ένα πολύ καλό κατάλογο εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι Ευρωπαίοι έτσι ώστε να υπεραμεινθούμε των αξιών μας. Και κυρίες και κύριοι, Και κυρίες και κύριοι πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση όπου στις κομματικές οικογένειες της Ευρώπης ε, το αίμα είναι πιο πυκνό από το νερό. Και τι γίνεται, αυτό σημαίνει ότι περασπίζονται τα μαύρα πρόβατα μέσα στις πολιτικές τους οικογένειες. Αν δείτε την έκθεση τα εκεί υπάρχουν τα εργαλεία. Πρόεδρος, ε, συνάδελφε κύριε Κονπεντήτη. Συνάδελφε Κονμπεντίτ, σας επιπλήτω για μια έκφραση που δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εδώ σε αυτή την αίθουσα και ο τελευταίος θα του δώσω το λόγο είναι ο κύριος Γκόλνης. Κύριε Πρόεδρε, μέχρι τώρα είχα την αίσθηση ότι οι ευρωπαϊκές αξίες ε, περιελάμβαναν και το σεβασμό του πληραλισμού, την αντιπαράθεση των ιδεών,